συνάδελφοι, τη συνεδρίαση της 5η 12ης ε, Μαρτίου. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις, έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά. Όχι. Δεν υπάρχουν ενστάσει. Ωραία, λοιπόν, έγκριναν τα πρακτικά. Να σα ανακοινώσω ότι ο κ. Βάλτης ε, διορίστηκε λετωνό